Ας συνεχίσουμε λοιπόν την σύνοδό μας. Τα πρακτικά της θεσινής συνεδριάσεως ε, είναι στη διάθεσή σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω όσον αφορά το σημείο 16 των πρακτικών. Το σημείο 16 των πρακτικών, σωστά, υπενθυμίζει ότι ζήτησα μια συζήτηση να ξεκινήσει όσον αφορά την άρση της κοινοβουλευτικής μου και την αρνηθήκατε. Αυτό είναι αντίθετο με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως από την κυρία Πρόεδρο Αντζελίλη που προείδρευε τη Συνόδου που ισχυρίστηκε ότι έλαβα το λόγο χθες όσον αφορά την άρση κοινοβουλευτική μου ασυλίας κάτι που είναι ψευδές. Το Κοινοβούλιο με στέρισε στέλνει από την προστασία αυτή ένα από τα μέλη του χωρίς να μπορέσει κανείς να τοποθετηθεί από αυτού στην Ολομέλεια ούτε ενδιαφερόμενο, ούτε εκείνο που θα μπορούσε να τον υπερασπιστεί, ούτε συζήτηση έγινε, ούτε επεξήγηση ψήφου, οτιδήποτε ήθελα αυτό να ε, καταγραφεί, να καταχωρηθεί και να σημειωθεί και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Πρόκειται περί παρατηρήσεών σας που αφορούν τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης.